Eh, Αγαπητοί συνάδελφοι, κηρύσω την επανέναρξη της ε, Συνόδου Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που διακόπη στις 13 Φεβρουαρίου. Καλώ τους ε, βουλευτές, επειδή δεν θα γίνει, επειδή δεν έχουμε και πάρα πολύ κόσμο παρόντα, να αραιώσετε λίγο, ε, ώστε να αραιώσετε, να μην κάθεστε δίπλα-δίπλα ένα στον άλλο για προφανείς υγειονομικούς λόγους. Ε, για τα πρακτικά της 13ης Φεβρουαρίου τα εγκεκριμένα κείμενα έχουν ήδη διανεμηθεί. Υπάρχουν παρατηρήσεις. Εάν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις, ε, τα, θεωρείται πως εγκρίνονται τα πρακτικά. Κάποιες ανακοινώσεις μετά από την εκλογή του κυρίου Ματ Κάρτι, ε, βουλευτή στο Εθνικό Κοινοβούλιο της Ιρλανδίας. Το Κοινοβούλιο διαπιστώνει την ε, κένωση της έδρας του ε, που τρέχει από τις 8 Φεβρουαρίου 2020 σύμφωνα με τον ιστορικό μας κανονισμό. Οι αρμόδιες αρχές της Ιρλανδίας μου την εκλογή στο Ευρωκοινοβουλίο του κυρίου Κρίς Μακμάνους ε, που θα αντικαταστήσει τον κύριο Ματ Κάρθι από τις 6 Μαρτίου 2020. Καλωσορίζουμε τον νέο συνάδελφο και ε, θυμίζω ότι θα αναλάβει τα καθήκοντά του σύμφωνα με τα όσα προβλέπει ο ιστορικός μας κανονισμός. Οι ομάδες S&D Renew και οι Πράσινοι μου ανακοίνωσαν ορισμένες αποφάσεις τροποποίησης σε σχέση με τους διορισμούς στις επιτροπές και τις αντιπροσωπείες. Οι αποφάσεις αυτές θα περιληφθούν στα πρακτικά της σημερινής συνεδρίασης και θα αρχίσουν να ισχύουν από τη σημερινή ε, ημερομηνία. Οι πρόεδροι των, επιτρο... των αρμοδίων επιτροπών ε, δεν έλαβαν αντιρρήσει ε, για τη σύσταση τη Επιτροπής Άγκρη να μην αντισταθούν σε κατεξοδότηση πράξη σύμφωνα με το άρθρο 111 παράγραφος 6 του κανονισμού. Η σύσταση είναι διαθέσιμη στο site της Ολομέλειας. Ε, αν μετά από 24 ώρες από την ανακοίνωση καμία πολιτική ομάδα ή ε, ικανός βουλευτών δεν γύρει θα θεωρηθεί πω εκρίνεται αυτή η σύσταση. Σε αντίθετη περίπτωση, θα τεθεί σε ψηφοφορία. Περνάμε τώρα στην ημερήσια διάταξη. Αγαπητοί συνάδελφοι, όπως σας ανακοίνωσα την περασμένη Πέμπτη, η συνεδρίαση της Ολομέλειας αυτή την εβδομάδα θα γίνει κατ' εξαίρεση εδώ στις Βρυξέλλες λόγω ανωτέρας βίας. Έλαβα αυτή την απόφαση επί τη βάση της έκθεσης της ιατρικής υπηρεσίας του Κοινοβουλίου, το οποίο μετά από ενδελεχή ανάλυση της εξέλιξης της επιδημίας του ιού COVID-19 του κορώνα ιού, ε, <coughs> θεώρησε πως η μετακίνηση του Ευρωκοινοβουλίου προς το Στρασβούργο για την ε, τέλεση της Ολομέλειας εκεί αποτελούσε σημαντικά ψηλότερο κίνδυνο για την υγεία μας για την υγεία και για την υγεία του τοπικού πληθυσμού. Ε, διαπιστώσαμε λοιπόν και δεχτήκαμε ότι δεν υπάρχουν πια οι απαραίτητες συνθήκες για να εγγυηθούμε την ασφάλεια όλων των συμμετεχόντων στην Ολομέλεια. Η απόφαση λοιπόν να γίνει η Ολομέλεια εδώ στις Βρυξέλλες ελήφθη στο πνεύμα και με πρόθεση να δοθεί συνέχεια στις εργασίες του Κοινοβουλίου και να μην διακοπούν οι ε, νομοθετικές δραστηριότητες. Θέλω να ευχαριστήσω τις γαλλικές αρχές και όσους ε, συμμετείχαν σε αυτή τη διαδικασία για την συνεργασία τους. Να ευχαριστήσω δε και το διοικητικό μηχανισμό του Κοινοβουλίου που εδώ και εβδομάδες παρακολουθεί τις εξελίξεις. Ζούμε μια δύσκολη στιγμή για το θεσμό μας και πρέπει να είναι καθήκον όλων μας, όλων των, βουλευτών, όλων των πολιτικών ομάδων να προστατευθεί η, ε, η βουλευτική δραστηριότητα για να μπορέσει να συνεχιστεί η δημοκρατική μας ζωή. Οι κυβερνήσεις μας και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητούν θυσίες από τους πολίτες μας και εμείς καλούμεθα να δώσουμε το καλό παράδειγμα. Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε όσο περισσότερο μπορούμε ώστε να εξασφαλίσουμε τη συνέχεια της ζωής και της ε, νομοπαραγωγικής διαδικασίας και του προϋπολογισμού. Η απόφαση λοιπόν για να καταπολεμηθεί ο COVID-19 να διατηρηθούν οι θέσεις απασχόλησης η οικονομία μας η οποία πλήττεται πολύ σκληρά αυτή τη στιγμή αλλά και για να συνεχίσουμε τις εργασίες μας για το Πράσινο Σύμφωνο, για τη μετανάστευση, για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Όλα αυτά μας επιβάλλουν να μείνουμε στις επάλξεις. Η σκέψη μας βέβαια πάει αυτή τη στιγμή σε όλους τους συναδέλφους που βρίσκονται στις ε, κόκκινες ζώνες και δεν μπορούν να κινηθούν. Για να είναι και εκείνοι στις ίδιες συνθήκες σας καλώ να ακολουθήσουμε τις συστάσεις των αρχών και ταυτόχρονα να εξετάσουμε τη πιθανότητα σε αυτή τη φάση να παραμείνουμε στις Βρυξέλλες ώστε να, μειωθεί στο ελάχιστο, να μειωθούν στο ελάχιστο οι μετακινήσεις. Και ξέρουμε ότι οι μετακινήσεις όπως μπορέσαμε εξάλλου να το διαπιστώσουμε από τις επαληθεύσεις που κάναμε, είναι ένας λόγος ανησυχίας. Πρέπει λοιπόν να τιμήσουμε την ε, κοινοβουλευτική μας εντολή, να τιμήσουμε όσους στην Ευρώπη και στον κόσμο ε, κάνουν το καθήκον τους ε, καθημερινά για να περιορίσουν την εξάπλωση αυτής της ε, ασθένειας. Είμαι επιπισμένος πως με ευθύνη και περηφάνεια θα είμαστε στο ύψος αυτής της περίστασης. Για αυτούς τους λόγους σήμερα συγκάλεσα μια έκτακτη συνεδρίαση της διάσκεψης των Προέδρων και ευχαριστώ όλους για τη συνεργασία, για το πνεύμα το ανοιχτό που με το οποίο συμμετείχαν. Αποφασίσαμε να τροποποιήσουμε το σχέδιο το οριστικό της ημερήσιας διάταξης ε, αυτής της συνόδου ως εξής. Η Σύνοδος του Μαρτίου θα ε, είναι μόνο η αυριανή μέρα, 10 Μαρτίου και θα έχει ως εξή 9 με 12 δηλώσεις Συμβουλίου και Επιτροπής για την επιδημία κορώνα ιού και βεβαίως θέλουμε το Κοινοβούλιο να είναι παρόν και να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στον αγώνα κατά του ιού. Το απόγευμα 3 με 6 θα γίνουν δηλώσεις Συμβουλίου και Επιτροπής για τα πορίσματα της έκτακτης συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και ξέρουμε ότι στο Κοινοβούλιο το Κοινοβούλιο είναι ε, ε, παράγων σε αυτήν την υπόθεση. Θα ακολουθήσουν δηλώσεις, όπως είπα, ε, Συμβουλίου και Επιτροπής ε, για τη μετανάστευση και τα σύνορα Ελλάδας-Τουρκίας και την κοινή απάντηση που θέλει να δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτές οι αλλαγές εγκρίθηκαν από την διάσκεψη των Προέδρων και βεβαίως όπως όλοι καταλαβαίνουμε, θέλουμε το Κοινοβούλιο να μείνει ανοιχτό, λειτουργικό, αλλά φυσικά χρειάζεται να λάβουμε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις και να περιορίσουμε στο απολύτως απαραίτητο τις δραστηριότητε μας. Γι' αυτό το λόγο η... τώρα θα διακοπεί η συνεδρίαση και αύριο θα ξαναρχίσουν οι εργασίες μας στις 9 το πρωί. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία σας.